Λοιπόν, θεωρούμε ότι κρίθη όπως έχει μείνει σε διάταξη. Ευχαριστώ. Μία ανακοίνωση. Την ερχόμενη εβδομάδα θα συνεδριάσουμε στις 7 στο Στρασβούργο. όπου θα συναντηθούμε με μία αντιπροσωπεία και θα συζητήσουμε του Αμερικανικού Κογκρέσου για διάφορα θέματα και κυρίως για θέματα που αφορούν τη Συρία και το Ιράν και την Ινδία. Νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα σκόπιμο. Και κατόπιν θα υπάρξει μια σύντομη δεξίωση, όπου θα έρθει και η κυρία Άστον. Θα ήθελα παρακαλώ ώστε να τον περισσότεροι να αξιοποιήσουν αυτή την ευκαιρία να κάνουμε αυτή την ανταλλαγή απόψεων. Επίσης, η προθεσμία για την γνωμοδότηση της κυρίας Ρομέρο Λόπεθ είναι η 18η Ιουνίου μεσημέρι. Απόγευμα ας πούμε. Γιατί είναι και Δευτέρα. Ε, διότι ξέρετε ότι οι υπάλληλοι θα είναι βεβαίω εδώ αλλά οι βουλευτές είναι ακόμη ε, καθοδόν. Εντάξει, συμφωνούμε. 18, 6 ώρα το απόγευμα. Ας περάσουμε τώρα στα πρακτικά. Ευρωπαϊκή Ένωση Ισραήλ νομίζω ότι υπήρξε τις τελευταίες μέρες ανταλλαγή απόψεων, υπήρξαν συμβαστικές τροπολογίες Δεν ξέρω ποιο θα μα ανακοινώσει τι έγινε. Στην τελευταία συνεδρίαση αποφασίστηκε να αναβληθεί η ψηφοφορία μέχρι την συνεδρίαση του ε, Ιουνίου για να διευκρινιστούν ε, διάφορα ε, σημεία όσον αφορά την πεδίο εφαρμογή. Το ζήτησε ο, Επίτρο, ο Επίτροπο κ. Ντεχούχτ. Αποστήλαμε επιστολή στον κ. Ντεχούχτ και τον κ. Μορέλη για να, μας, να πούμε τι πρέπει να διευκρινίσει η Επιτροπή, με βάση το έγγραφο και τις νομικές μας υπηρεσίες, η Επιτροπή μας ενημέρωσε η Επιτροπή μας ενημέρωσε ότι δεν μπορούσε να μας στείλει αυτή ε, τη διευκρίνηση πριν την 7η Ιουνίου, διότι πρέπει να συμφωνήσει συνολικά το Σώμα των Επιτρόπων και γι' αυτό χρειάζεται και νομική εμπειρογνώμηση. Η κυρία Ντεκάιζερ συζήτησε το συμβαστικό κείμενο με τους, συναδρές, με συναδέλφους από διάφορες πολιτικές ομάδες και με τους σκιώδεις ηγητές για να αντικατοπτρίζει τη σημερινή κατάσταση και ίσως θα ήταν δυνατόν η ίντα με τις προτάσεις που έκανε στο γράμμα θα υποβάλει προφορική ερώτηση στην Ολομέλεια. Θα μπορούσαμε λοιπόν και εμείς να ε, συμμετάσχουμε σε αυτή την προφορική ερώτηση. Αλλά δεν με ικανοποιεί ούτε η συμπεριφορά της Επιτροπής, ούτε ε, ο τρόπος με τον οποίο χρονοτριβούν. Θα έπρεπε να το έχουν πει από την αρχή. Στην αρχή να λένε ότι είναι επίγον, μετά να λένε είναι αρκετά επίγον και τώρα να δημιουργηθούν ε, θέματα καθυστέρησης. Βεβαίως ε, υπάρχουν θέματα πρωτοκόλου, αλλά αυτά μπορεί να φύλλονται σε πολιτικούς λόγους, στους οποίους δεν θα αναφερθώ δημοσίω, αλλά δεν είναι τρόπος αυτός να αντιμετωπίζουμε τα θέματα και γι' αυτό θεωρώ ότι την επόμενη φορά θα πρέπει να το χειριστούμε διαφορετικά. Η Επιτροπή θα πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν μπορούν να παίζουν τέτοια παιχνίδια. Η κυρία Ντε Κέζερ. Παρακαλώ. Χωρίς μικρόφωνο. Χωρίς μικρόφωνο. Ευχαριστώ. Όπως είπατε και στην προηγούμενη συνεδρίασή μας αφέτ για το θέμα αυτό, στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει προχωρήσει το θέμα εφόσον καταλήγουν σήμερα σε ένα συμβιβασμό που βεβαίως δεν ικανοποιεί καμία πολιτική ομάδα ούτε τη δική μου αλλά είναι ένα συμβασμός α, τον οποίο μπορούμε να δεχθούμε και νομίζω ότι θα ηρεμήσει τα πράγματα για αυτό το τόσο ευαίσθητο θέμα. Ευχαριστώ όλους τους σκιώδεις και θα έλεγα και εσάς βεβαίως κύριε Πρόεδρε για την ε, ιδιαίτερη κατανόηση που επιδείξατε για το θέμα αυτό και ο μου ε, και τον συνάδελφό μου Σαλαφράγκα θέλω να ευχαριστήσω που έπαιξε το ρόλο διαμεσολαβητή. Πιστεύω ότι ο συμβασμό που πιστεύω ότι είναι λοιπόν αποδεκτός και στην Επιτροπή μας, αλλά όχι μόνο. Θα μπορούσε να τον δεχθεί και η Ίντα που θα αναλάβει τη σκητάλη μετά από εμά. Σας καλώ λοιπόν θερμός να συμφωνήσετε με τη συμβαστική άποψη και την έκθεση. Η Επιτροπή ΑΦΕΤ διαβάζω καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου που είναι η επί της αρμόδια να συνενέσει είναι σημαντικός πιστεύω όρος να συνενέσει στο πρωτόκολλο αυτό εφόσον οι νομικές προϋποθέσεις που αναφέρονται από τον πρόεδρο της ΑΦΕΤ, κύριο Έλμαρ Μπροκ, στον ε, ε, κύριο Κάρερ Ντεχούκτ, επίτροπο για το εμπόριο, εφόσον λοιπόν οι συνθήκες αυτές πληρούνται. Και βεβαίως θα επισυνάψουμε και την επιστολή που έστειλε ο κύριος Μπροκ στον κύριο Ντεχούκτ, που περιλαμβάνει τρία σημαντικά σημεία. Πρώτον, ο πρόεδρος της ΑΦΕΤ ζητάει νομικά δεσμευτικές διαβεβαιώσεις όσον αφορά την εδαφική αρμοδιότητα που αφορούν την αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 9 του πρωτοκόλλου ζητάει κανένα βιομηχανικό προϊόν που παράγεται στις, στους ε, ε, Ισραηλινούς επικισμούς στην Δυτική Όχθη ε, και τα βιομηχανικά προϊόντα που παράγονται στις ε, κατεχόμενες περιοχές με εξαίρεση αυτά που παράγονται στους επικισμούς να συμπεριλαμβάνονται, να αντιμετωπίζονται ισότιμα, με συγχωρείτε, οποιαδήποτε άλλα βιομηχανικά προϊόντα στα πλαίσια, στο πεδίο εφαρμογής αυτού του πρωτοκόλου. Αυτά αναφέρονταν στην επιστολή. Πρέπει λοιπόν η ίντα να ζητήσει διευκρινήσεις για τα σημεία αυτά, να ζητήσει να πληρούνται αυτές οι συνθήκες, είναι ακριβώς στο γράμμα των συνθήκων και ακριβώς σύμφωνα με μια ευρωπαϊκή πολιτική που επανειλημμένα έχει επιβεβαιωθεί. Η δημιουργία όλων αυτών των νομικά δεσμευτικών μηχανισμών μπορεί να γίνει στη διαδικασία εφαρμογής του πρωτοκόλου. Δεν ζητάμε εκ νέου διαπραγματεύσεις με τους Ισραηλινούς εταίρους. Όχι λοιπόν αναδιαπραγμάτευση του πρωτοκόλου και υπενθυμίζω ότι το πρωτόκολλο αυτό που αυτή τη στιγμή αφορά τα φαρμακευτικά προϊόντα ανοίξαμε τις συζητήσεις για το φαρμακευτικό τομέα στο εν λόγω παράρτημα μετά λοιπόν μπορεί να περάσουμε και σε άλλους τομείς όπου δεν χρειάζεται πλέον η γνώμη του Κοινοβουλίου. Άρα οι νομικά δεσμευτικές ε, αυτές προϋποθέσεις πρέπει να ισχύουν για οποιαδήποτε άλλα προϊόντα επίσης. Δεν ζητάμε επίσης από το Ισραήλ να παραβιάσει τους νόμους του. Δεν υποχρεωμένο να πει ότι δεν θεωρεί ότι τα προϊόντα από τους επικισμούς είναι από, αυτές, από αυτά τα εδάφη τις κατεχόμενες περιοχές, αλλά πρέπει να μας πει ότι δεν μπορεί να πιστοποιήσει τα προϊόντα από τους επικισμούς γιατί δεν τους αναγνωρίζουμε. Αυτό αποφασίστηκε, έγινε δεκτό και από μας, διότι θεωρούμε ότι είναι σύμφωνο με το πνεύμα και την ευρωπαϊκή πολιτική για την περιοχή αυτή, σεβόμενη βεβαίως τις ευαισθησίες των μεν και των δε. Σας καλώ λοιπόν να ψηφίσουμε. Θα ηρεμήσει τις συζητήσεις μας και θα επιτρέψει να διεξάγεται το εμπόριό μας με το Ισραήλ με βάση την ευρωπαϊκή μας πολιτική που αφορά την επίλυση μέσω δύο κρατών στα σύνορα του 67. Τα λέω όλα αυτά. Ευχαριστώ τους πάντες. Ήταν ιδιαίτερα δύσκολο και περίπλοκο το θέμα αυτό, αλλά παρόλα αυτά καταλήξαμε σε μια λύση αποδεκτή και καταδεικνύει την οριμότητα της Επιτροπής μας. Ο κύριος Τάνου. Ευχαριστώ. Η ομάδα μου δεν θα στηρίξει το συμβιβασμό αυτό, γιατί πιστεύουμε ότι είναι μια πολιτική χειρονομία. Δέχομαι βέβαια ότι μπορεί να επιτυχάνονται οι παρετέρω στόχοι μα και να μπορεί να υπάρξει συνένεση. Από την άλλη όμω είναι σαφέ για όλου μα, ότι προσπαθεί να κάνει σύνδεση με την τεχνική πιστοποίηση βιομηχανικών και άλλων προϊόντων, που είναι ένα τεράστιο θέμα που δεν έχει καμιά σχέση με την επίθεση που γίνεται στο Ισραήλ στα πλαίσια της επίλυσης. Δεν νομίζω λοιπόν ότι μπορεί να βοηθήσει. Από όσο ξέρω εγώ δεν υπάρχει παραγωγή τέτοιων προϊόντων. Οπότε νομίζω ότι εδώ πέρα μπαίνουμε σε μια εντελώ διαφορετική συζήτηση από ότι το τεχνικό ζήτημα που είναι η πιστοποίηση και δεν έχει να κάνει ούτε με την δαφικότητα από που προέρχονται τα προϊόντα αυτά. Απλώ δίνει δικαιώματα στι αρμόδιε αρχέ του Ισραήλ να πιστοποιούν ένα αγαθόν που είναι ικανοποιητικό για να κυκλοφορήσει προς κατανάλωση στην ε, Ευρώπη, όπως για παράδειγμα τα φάρμακα. Οπότε αυτό που κάνουμε είναι ότι τελικά τιμωρούμε τους πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ντροπή, ειλικρινά. Θα καταψηφίσουμε το συμβιβασμό, αλλά ελπίζω τελικά να περάσει και να λυθεί ικανοποιητικά για όλες τις πλευρές το ζήτημα. Ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε, γιατί λέτε Ευρωπαίοι και Βρετανοί καταναλωτέ, δεν είναι Ευρωπαίοι Βρετανοί καταναλωτέ. Ίσως κάποιοι στη χώρα μου να λέγανε πως όχι, αλλά... Και αυτό όμως είναι ένα θέμα, το πώς ε, καταλαβαίνει κανείς τα θέματα του, το τι είναι νομικά σωστό αυτό που είπατε και εσείς για τα φαρμακευτικά προϊόντα. Η κυρία Γιαννάκου, η Μαριέτα. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα αποδέχεται τον συνδυασμό ο οποίος έγινε μετά από πολλές συζητήσεις παρά το γεγονός ότι εμείς από την αρχή είχαμε τοποθετηθεί θετικά και θέλαμε να τελειώνει ε, σύντομα αυτή η υπόθεση. Νομίζω ότι η γνώμη αυτή που θα δώσουμε στην ε, ίντα μπορεί να εκφράσει και το γενικότερο αίσθημα της Επιτροπής και να διευκολύνει και τη συνεργασία εν συνεχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με το κράτος του Ισραήλ. Και θεωρώ ότι πρέπει να ψηφίσουμε κατευθείαν. Δεν βλέπω να θέλει κανείς άλλο το λόγο, τότε μπορούμε να βράσουμε στην ψηφοφορία. Ποιο είναι υπέρ τη συμβαστική τροπολογία 1. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται με πέντε ψήφους κατά. Τώρα ψηφοφορία. Α, πρέπει να κάνουμε και τώρα τελική ψηφοφορία. Ωραία, θα είναι ηλεκτρονική. Ποιοι είναι υπέρ αυτή τη νομοδότησης συνολικά παρακαλώ. Ο κύριος Σούλτ δεν έχει την κάρτα του. Εντάξει. Ωραία. Ψηφίζουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 41 υπέρ. Κύριε Σούλτ θέλετε να ψηφίσετε. Α, 42 υπέρ. 2 κατά 3 αποχές. Βεβαίω θα το παρακολουθήσουμε και τι επόμενε εβδομάδε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και την κυρία εισηγήτρια. Ευχαριστώ. Meine Damen und Herren. Κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε τώρα στην ανταλλαγή απόψεων για, την, για το εταιρικό όργανο για, σε σχέση με τις τρίτες χώρες. Χαιρετίζω τους εμπειρογνώμονες που έχουμε στη διάθεσή μας. Ο εισηγητής μας, κύριος Μάριο Μάουρο, είναι στην Οικονομική Επιτροπή σε μια ψηφοφορία αλλά βλέπω ότι τελειώσανε και είναι εδώ παρόν και δίνω το λόγο στον κύριο Μάριο Μάουρο. Όταν ένα σταλός πηγαίνει σε μια θέση στο κέντρο είναι επικίνδυνο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση. Οφείλεται στην ψηφοφορία στην Επιτροπή ΕΚΟΝ. Θα ήθελα και εγώ να καλωσορίσω τους ε, φιλοξενούμενους μας και να τους ευχαριστήσω που ήρθαν ε, για να πάρουν το λόγο στην Επιτροπή μας. Εγώ θεώρησα ότι ήταν σημαντικό να ζητήσουμε την διοργάνωση μιας περαιτέρω ανταλλαγή απόψεων για το μέσο εταιρική σχέσης γιατί θεωρώ πως είναι σκόπιμο να καλέσουμε την Κομισιόν, την, ε, την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να μας πούν την γνώμη τους όσον αφορά αυτό το μέσο εταιρική σχέσης και τον ε, στρατηγικό ρόλο που μπορεί να παίξει αυτό το μέσο στο πλαίσιο των εξωτερικών σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεωρώ λοιπόν ότι υπάρχουν επιτυχίες στην πρόταση της Κομισιόν που απαιτούν αποσαφήνιση ε, ή εμβάθυνση. Θα ήθελα να θυμίσω λοιπόν στους φιλοξενούμενους μας ότι σήμερα είναι η ευκαιρία για να ξεκινήσουμε ένα κοινό προβληματισμό για το ποια είναι τα στοιχεία που μπορούν να ενισχύσουν το πεδίο το του μέσου αυτού και να καταστήσουν αυτό το μέσο πιο επίκαιρο και πιο αποτελεσματικό στην απόδοσή του. Επίσης θα ήθελα να τονίσω τη σημασία μιας πλήρους κατανόησης από πλευράς των Ευρωπαίων πολιτών όσον αφορά τους στόχους αυτού του μέσου εταιρικής σχέσης. Το ερώτημα λοιπόν που απευθύνω σε όλους μας τους ε, καλεσμένους και που ελπίζω να θα μπορέσουν να τα απαντήσουν στη διάρκεια της συζήτησης είναι το εξή. Γνωρίζουμε ότι το μέσο εταιρική σχέση είναι ένα μέσο εξωτερικής πολιτικής που στόχο έχει να χρηματοδοτεί τις διμερείς σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιες είναι ωστόσο οι συγκεκριμένες δραστηριότητες που μπορούν ε, να εξεταστούν τα προγράμματα και τα, οι στόχοι που θα επιδιωχθούν χάρη στο μέσο εταιρική σχέση. Η ταυτότητα αυτού του μέσου, κατά τη γνώμη μου, είναι καθαρά εξωτερική πολιτική. Αλλά ποια είναι η βασική οπτική, ποια είναι τα στρατηγικά συμφέροντα τη Ένωση που θέλουμε εμεί έτσι να προωθήσουμε. Η πρόταση της Κομισιόν επίσης διατυπώνει κάποιες προτάσεις, ε, όχι αποκλειστικού τύπου, στο παράρτημα. Αλλά πρόκειται για κάποιες γενικόλογες δηλώσεις που είναι κάπως υπερβολικές και όχι στρατηγικού χαρακτήρα όσον αφορά μελέτες και ερευνητικά προγράμματα. Εγώ θέλω να είμαι ακόμα πιο σαφής. Είναι προφανές ότι είναι σημαντικές δραστηριότητες, αλλά δεν μπορούν αυτές να παίζουν τον κεντρικό ρόλο. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να προσδώσουμε στο παράρτημα ένα πολύ πιο προγραμματικό χαρακτήρα που θα εντοπίζει ξεκάθαρες κατευθυντήριες γραμμές για τη χρήση των διαθέσιμων πόρων επί τη βάση του μέσου της, της εταιρικής σχέσης. Ποια είναι λοιπόν η στήριξη που θα προσφέρει αυτό το μέσο στην εξωτερική πολιτική ε, της Ένωσης. Ποια είναι η προστιθέμενη αξία που θέλει να δημιουργήσει στο πλαίσιο αυτής της εξωτερικής μας πολιτικής. Και έπειτα ακόμα ένα ερώτημα που θέλω να διατυπώσω. Σε αυτή την... Ε, αυτό το ερώτημα είναι μόνο για την Κομισιόν και για την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και το Συμβούλιο. Το άρθρο 5, παράγραφος 5 της πρότασης της Κομισιόν προβλέπει τη δυνατότητα δημιουργίας ενός αποθεματικού για τα κονδύλια που δεν έχουν ε, χορηγηθεί σε συγκεκριμένα προγράμματα. Γιατί προβλέπετε μόνο στο μέσο εταιρική σχέση αυτό το αποθεματικό, πώς θα λειτουργήσει, ποιο ποσοστό θα ε, περιλαμβάνεται και ποια θα είναι η διαδικασία για την καταχώρηση των κονδυλίων στο αποθεματικό. Και τέλος μια τελευταία ερώτηση που απευθύνω στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Με ποιο τρόπο, κατά τη γνώμη σας, τα κονδύλια του μέσου εταιρική σχέση θα μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν ως εγγύηση για δάνεια από την ε, Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων σε σχέση με χώρες που είναι εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για παράδειγμα, για να υλοποιηθούν στόχοι της, της, Στρατηγικής Ευρώπη 2020. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Να, τώρα ο κύριος Αντρικίνικεμ που είναι ο εισηγητής της ΣΥΝΤΑ. Η κυρία, συγγνώμη. Ευχαριστώ. Είμαι η συγκήτρια από την ΙΝΤΕ και την γνωμοδότησή της. Βάσει του άρθρου 50 λοιπόν του κανονισμού υποβάλλεται η γνωμοδότηση αυτή που σημαίνει ότι συνεισφέρει η Επιτροπή μας και στα Το μέσο αυτοτερικής σχέσης σκοπεύει στη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες εκείνες οι οποίες μπορούν να αποφελθούν από διμερή ε, βοήθεια. Κίνα, Ρωσία, χώρες Λατινικής Αμερικής. Στόχος είναι να προωθήσει τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να αντιμετωπίσει παγκόσμιες προκλήσεις και να βοηθήσει στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής του 2020. Είναι ένα οικονομικό μέσο για τη συνεργασία με τις εκβιομηχανισμένε και λοιπές υψηλού εισοδήματο χώρες και εδάφη. Είχαμε το ICI λοιπόν, το μέσο αυτό, μέχρι να πάρει τη σκητάλη το μέσο εταιρική σχέση. Θέλουμε κάποιε διευκρινήσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όμω για κάποια συγκεκριμένα ζητήματα. Τι υποβάλαμε, αλλά απαντήσει δεν έχουμε πάρει ακόμα. Πρώτον, η στόχη κλειδί του μέσου είναι η βελτίωση της πρόσβασης στις αγορές και αναπτυσσόμενο εμπόριο. Εμεί ε, πιστεύουμε ότι η στρατηγική τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την προώθηση τη οικονομική συνεργασίας και του εμπορίου πρέπει να βασίζεται σε μια ανάλυση σε βάθο των τάσεων που υπάρχουν στον κόσμο όσον αφορά το εμπόριο. Οπότε ρωτάω, η Επιτροπή μπορεί να μα εξηγήσει τι ακριβώ είναι αυτέ οι δραστηριότητε. Μπορεί να μα δώσει παραδείγματα η Επιτροπή για αντίστοιχε δραστηριότητε οι οποίε μέχρι τώρα έχουν χρηματοδοτηθεί. Και γιατί οι χώρε μιλάμε, ποιε περιφέρειε υποφελούνται από αυτέ ε, τι δράσει. Δεύτερον, τι προτερότητες έχουμε όσον αφορά τις χώρες και τις περιφέρειες, προκειμένου να πετύχουμε τους στόχους του σχετικούς με το εμπόριο. Τρίτον, στον κανονισμό η πρόταση προτείνει 20% ε, μη ουσιοδών τροποποίησεων όσον αφορά τα ετήσια διοικητικά προγράμματα. Οπότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να μας εξηγήσει ποια επιχειρήματα βρίσκονται πίσω από αυτό το 20%, γιατί 20% και όχι 10%. Η Επιτροπή λοιπόν μπορεί να μας πει προβλέπετε διαβούλευση ανάμεσα στην Επιτροπή και τα κράτη-μέλη, τους ζωρητές, τους διάφορους ε, φορείς, τους ενδιαφερόμενους, τις τοπικές αρχές, στην αρχή της διαδικασίας, προκειμένου να υπάρξει συμπληρωματικότητα και να έχουμε και τη συνεργασία των φορέων αυτών. Τέλος, Οι προτεραιότητες όσον αφορά τις περιφέρειες στρατηγικής σημασίας και περιφέρειες με τις οποίες συνεργαζόμαστε. Υπάρχει αξιολόγηση εξάντε όσον αφορά τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν αποφασιστούν τα αιτήσια διοικητικά προγράμματα. Έχει γίνει κάτι τέτοιο ή προβλέπεται μια τέτοια αξιολόγηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Να ξεκινήσουμε λοιπόν τη συζήτηση εμπειρογνώμονε, θα πάρουν το λόγο. Ο κύριος Τούγκλα Μαγκή. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ πολύ την Επιτροπή για τον τρόπο με τον οποίο έχετε αντιμετωπίσει το μέσο εταιρική σχέση, την προσοχή δηλαδή που του έχετε επιφυλάξει. Θέλουμε να εξηγήσουμε λοιπόν από τη δικιά μας την πλευρά πώς μπορεί να λειτουργήσει αυτό το μέσο και τι μπορεί να πετύχει. Εμείς το βλέπουμε σαν ένα μεγάλο καινοτόμο μέσο στις προτάσεις του πολιτικού δημοσιονομικού πλαισίου. Πρέπει να το δούμε σαν κάτι που μπορεί να πάει πολύ μακριά και που μπορεί να αντιμετωπίσει παγκόσμιες προκλήσεις όπως είναι οι κλιματικές αλλαγές αλλά και το ενεργειακό. Μπορεί επίσης να στηρίξει και την εξωτερική διάσταση της ευρωπαϊκής πολιτικής. Πολλές από τις τροπολογίες που προτείνει ο εισηγητής ενισχύουν τους στόχους μας αυτούς. Εμείς βλέπουμε ότι έχει δύο σκέλη. Πρώτα απ' όλα σε παγκόσμιο επίπεδο μπορούμε να διευρύνουμε τη συνεργασία μας, μπορούμε να έχουμε περισσότερες σχέσεις με χώρες οι οποίες είναι στρατηγική σημασία τέρη μας, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ιαπωνία αλλά και οι χώρες BRICS, αλλά από την άλλη μπορούμε έτσι να στηρίξουμε και κάθε είδους πολιτικού διαλόγου. Θα βοηθήσει επίση το μέσο αυτό να ενισχύσουμε και τι σχέσει μα με τι χώρε εκείνες οι οποίε δεν επιλέγονται στα πλαίσια τη αναπτυξιακή βοήθεια. Φυσικά θα πάρουμε τα μαθήματα που πρέπει από το ICI και το ICI-SIN. Έτσι λοιπόν θα μπορέσουμε να δουλέψουμε σε ευρύτερα πλαίσια με όλες τις χώρες οι οποίες καλύπτονται, αλλά θα μπορούμε να προβλέψουμε και άλλου είδους δραστηριότητες. Και αντίθετα με τα όσα συμβαίνουν με το ICI και το ICI-SIN, το μέσο αυτό θα πηγαίνει πιο μακριά, γιατί θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε οποιαδήποτε χώρα με την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ε, στρατηγικά συμφέροντα ή συμφέροντα τα οποία μπορούμε να προβλέψουμε ότι δημιουργούνται ad hoc. Υπάρχει και ευελιξία, η οποία θα επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ανταποκριθεί σε αλλαγές που συμβαίνουν με τις χώρες τέρους μας και θα μπορέσει επίσης να δράσει στην παγκόσμια σκηνή μέσα στις ε, αλλαγές οι οποίες συνεχώς λαμβάνουν χώρα. Δεν αναφέρονται συγκεκριμένε χώρε ή ομάδε χωρών, αλλά από πλευρά δραστηριοτήτων πρέπει να σα πω ότι ο στόχο μα είναι να αντιμετωπίσουμε μεγάλες προκλήσεις αλλά και άλλα αριθμιστικά ζητήματα ευρύτερα υπέρ της πολιτικής σταθερότητας, έτσι όπως προτείνει και ο εισηγητής. Προωθεί επίση τα συμφέροντα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ενισχύοντα την εξωτερική σχέση των ευρωπαϊκών πολιτικών. Ο κύριος Γκουγεντέο, συνάδελφό μου, θα σα δώσει περισσότερε λεπτομέρειε για αυτά τα στοιχεία σε λίγο. Επιπλέον, το μέσο εταιρική σχέση θα χρησιμοποιηθεί και για να ξεκινήσουν συγκεκριμένε πρωτοβουλίε όσον αφορά τον πολιτικό διάλογο μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και τρίτων χωρών. Θέλω εδώ να αναφέρω ότι ένα από του κύριου στόχου, όπω αναφέρει και η συγκέντρια τη ΣΥΝΤΑ, είναι να προσφέρει ένα ασφαλέ επενδυτικό πλαίσιο και να προσφέρει νέε ευκαιρίε στι ευρωπαϊκέ επιχειρήσει διεθνώ. Θέλω όμω να επιμείνω επίση και στο ότι θα αποτελεί το κύριο μέσο εξωτερικού προσανατολισμού για να πετύχουμε του στόχου μα πέρα από την αναπτυξιακή συνεργασία. Είναι κάτι το οποίο δεν είναι βοήθεια, δεν συνδέεται με την ανακούφιση από την φτώχεια. Μιλάμε εδώ πέρα περισσότερο για εταίρους και όχι για, για δικαιούχους. Είναι πάντως ένα θέμα πάνω στο οποίο πρέπει να παραμείνουμε ρεαλιστικοί για το ρόλο των κυβερνήσεων. Είναι ζωτική σημασία. Αν θέλουμε να τηρούνται οι ευρωπαϊκές προδιαγραφές και να πάψουν να υπάρχουν εμπορικά εμπόδια. Το πλαίσιο της κοινωνίας των πολιτών επίσης θα μας απασχολήσει στο διάλογο που θα έχουμε σε όλα τα επίπεδα ή και στα πλαίσια τι ε, διπλωματίε που θα χρησιμοποιήσουμε. Επιτρέψτε μου τώρα σύντομα να αναφερθώ και σε κάποια ζητήματα τα οποία εμεί πιστεύουμε ότι στην ε, έκθεση των εισηγητών μπορεί να δημιουργήσουν ε, κάποιες ανησυχίες επειδή υπάρχουν αποκλήσεις. Για τον αντίκτυπο. Λέτε ότι ο αντίκτυπος πρέπει να φαίνεται από τις αλλαγές και πρέπει να υπάρχει έλεγχος και αξιολόγηση βάσει προκαθορισμένων και σαφών δικτών. Εμείς συμφωνούμε μεν σε αυτό, ότι δηλαδή πρέπει να υπάρξει βελτίωση προς τη θέμενη αξία, αλλά πρέπει επίσης να λογοδοτούμε. Εμείς πιστεύουμε ότι μια τέτοια πρόταση για λεπτομερείς δείκτες που πρέπει εξάντε να καθοριστούν, είναι κάτι που δημιουργεί δυσκολίες για ορισμένους τομείς πολιτικής. Και μάλιστα μπορεί να εμποδίσει και τις δραστηριότητες και το έργο, γιατί φτάνουν ευρύτερες ε, συμφωνίες, διμερείς συμφωνίες ή δηλώσεις απλώς. Ένα άλλο θέμα είναι η ελαστικότητα. Ο συγητής προτείνει περιορισμένη ελαστικότητα και καθόλου. Αυτό όμως θα αποτελέσει εμπόδιο προκειμένου το μέσο αυτό να μπορέσει να ανταποκριθεί στις ανάγκες. Πρέπει να μπορούμε να δίνουμε απαντήσεις γρήγορα στις πολιτικές αλλαγές και να στηρίζουμε πολιτικούς στόχους με τους εταίρους μας. Τέλος, πιστεύουμε ότι το περιεχόμενο του παραρτήματος είναι πάρα πολύ ακριβές και λεπτομερές. Και εδώ πιστεύουμε ότι οι επιπλέον περιγραφές θα εμποδίσουν την λειτουργία του μέσου, γιατί σημαίνει ότι οποιαδήποτε δράση, οποιοδήποτε θεματικός τομέας, ο οποίος δεν υπογραμμίζεται συγκεκριμένα, αποκλείεται. Εμείς πιστεύουμε ότι κάτι τέτοιο πρέπει να μείνει στον ετήσιο σχεδιασμό. Να περιληφθεί εκεί. Πρόεδρε, είμαστε έτοιμοι να κοιτάξουμε συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν να προσθεθούν ώστε να έχουμε ένα πιο συγκεκριμένο και πιο εύκολα κατανοητό πλαίσιο. Εδώ θα σταματήσω, Πρόεδρε, και αν μου επιτρέπετε να δώσω το λόγο στον κύριο Γιλαντέ, ο οποίος θα μας παρουσιάσει περισσότερες λεπτομέρειες για τα άλλα σημαντικά στοιχεία του μέσου εταιρικής σχέσης. the floor has Daniel Gouillardet. Daniel Είναι υπεύθυνο για είναι ματάρχης για θέματα σφελικής συνεργασίας και αντιτρομοκρατική δραστηριότητα. θα μιλήσω κυρίως για τις σφαιρικές προκλήσεις για αυτό το μέσο εταιρική σχέσης. Να μιλήσω για μερικά μόνο στοιχεία, διότι η κυρία Άστον θέλησε να υπάρξει αυτό το μέσο, είναι ένα νέο εργαλείο στο κουτί με τα εργαλεία μας. Αφορούν μερικά συγκεκριμένα χώρα, μερικές συγκεκριμένες χώρες ενέργειες αυτές στο παρελθόν. Τώρα έχουμε ένα σφαιρικό μέσο καλύπτει όλη μας την προσπάθεια να υπάρξει διάλογος με όλες τις χώρες και με όλους τους τομείς. Μεγάλη αλλαγή σε σχέση με το παρελθόν. Τίποτα δεν είναι βέβαια τέλειο, αλλά τουλάχιστον τώρα υπάρχει αυτό το μέσο. Η πρόταση καλύτερα υπάρχει και ελπίζουμε να υπάρξει απόφαση. Είναι βεβαίως ε, κάτι που θα μας βοηθήσει στο μέλλον για να υπερασπιστούμε τα συμφέροντά μας στα πλαίσια του διαλόγου με τους στρατηγικούς μας εταίρους. Δεύτερον, προωθούμε έναντι τρίτων χωρών την ευρωπαϊκή πολιτική. Γι' αυτό ε, επικεντρωνόμεθα στη στρατηγική Ευρώπη 2020 με μερικές σημαντικές νέες πολιτικές, κλιματική αλλαγή, προστασία του περιβάλλοντος, και ενέργεια σε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι στοιχεία που ήδη τα συζητάμε με αρκετούς εταίρους στον κόσμο Οπότε το μέσο εταιρικής σχέσης θα, θα επιτρέψει στην Ένωση να έχει ένα μέσο συνεργασίας στη διάθεσή της που δεν είναι μόνο μέσο επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας αλλά και για δραστηριότητες που δεν είναι του τύπου της ε, δημόσιας αναπτυξιακής βοήθειας αλλά θα αφορά διάφορους τομείς όπου η συνεργασία είναι σημαντική. Συμφωνώ με αυτό που είπε ο προηγούμενος ομιλητής ότι το στοιχείο αυτό θα πρέπει να αναφέρεται συγκεκριμένα στον κανονισμό που εξετάζεται. Θέλουμε λοιπόν να υπάρχει συνεργασία, κοινή δράση στις ενέργειες που αφορούν τον τομέα αυτό και ιδιαίτερα στους τομείς εμπορίου που ανέφερε και ο εισηγητής Ίντα. Προωθούμε λοιπόν εμπορικές δραστηριότητες μέσω του εμπορικού διαλόγου που θα διεξάγεται στα πλαίσια αυτής της συμφωνίας. Υπάρχει λοιπόν πολιτικό πλαίσιο για τις συμφωνίες που έχουμε με πολλές χώρες, με πολλούς στρατηγικούς εταίρους πιο συγκεκριμένα και θα υπάρχει ένα μέσο για να μας βοηθήσει πέρα από την παραδοσιακή αναπτυξιακή συνεργασία και τα μέσα για αυτήν την αναπτυξιακή συνεργασία που είχαμε και στο παρελθόν. Ορίστε λοιπόν σημαντικά στοιχεία για το πεδίο εφαρμογής, την ευελιξία και την επίπτωση στις ε, σχέσεις μας με τις χώρες αυτές εταίρους μας. Η συνάδελφος ε, Έλλης Μάθιους θα πει περισσότερα για το πώς αυτό το μέσο θα συνδυαστεί με τον πολιτικό και τομεακό διάλογο με συγκεκριμένε χώρες και έχουμε και μερικά παραδείγματα. Ελίζα, έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Α, συγγνώμη, ο κύριος Έλλη Μάθιος. Αναπληρωτής τμήματάρχη για σχέσεις με Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά. Σας ευχαριστώ πολύ. Όπως, όπως ήδη είπατε, είμαι από, προέρχομαι από το τμήμα σχέσεων με τη ΣΥΠΑ και τον Καναδά και είμαστε ένα από τα βασικά τμήματα που θα αναμειχθούμε στην ανάπτυξη αυτού του μέσου. Όπως είπε ο συνάδελφος, εγώ πιστεύω ότι όπως το προτείναμε αυτό το μέσο, βασικά θέλουμε να στηρίξουμε τις στρατηγικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βασικά με τους στρατηγικούς εταίρους όπως αυτοί αποκαλούνται, αλλά Επίση, όπω αναφέρθηκε και σε άλλε επιτροπέ, με άλλε χώρε που έχουμε επίση στρατηγικά συμφέροντα, αλλά που δεν εντάσσονται επισήμω στου στρατηγικού μα εταίρου. Αυτό που θα ήθελα να κάνω είναι να σας δώσω κάποια παραδείγματα για τα πράγματα που θα μπορούσε να στηρίξει το μέσο εταιρικής σχέσης. Ε, απλά ενδεικτικά σας τα αναφέρω. Αυτό το τονίζω, αλλά στόχο έχουν να δείξουν με ποιο τρόπο θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε κάποια από τα ζητήματα που προέκυψαν μέσα από τις λεπτομερείς προτάσεις τροπολογίας που έχει υποβάλει η εισηγητής όσον αφορά το παράρτημα. Και θα επιλέξω τρεις χώρες σημαντικές ε, Βραζιλία, Κίνα και Ινδία. Για παράδειγμα, με τη Βραζιλία θα μπορούσαμε να στηρίξουμε ειδικέ ε, πτυχές του διαλόγου πολιτικής για τις κλιματικές αλλαγέ ε, συμπεριλαμβανομένων μηχανισμών της αγοράς, να δουλέψουμε για δραστηριότητε που θα ανέπτυσαν περισσότερο τη συνεργασία μας στο διάστημα και στην πλοήγηση δορυφόρων. Επίσης, θα μπορούσαμε να στηρίξουμε σε ένα άλλο παράδειγμα αριθμιστικό διάλογο στον τομέα των ε, προϊόντων ξυλία, ε, δασοκομεία ή σε τομέα των ορυκτών. Όλα αυτά είναι ε, υλικά τα οποία περιλαμβάνονται και στι προτάσει τροπολογιών του ίδιου του εισηγητή. Με την Κίνα και πάλι, απλά ενδεικτικά σα λέω ότι θα μπορούσαμε να στηρίξουμε δραστηριότητε, να προωθήσουμε δραστηριότητε που στηρίζουν την εταιρική σχέση για την αστικοποίηση. Επίσης θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε την Κίνα να δει και να εξετάσει το σύστημα ανταλλαγή εκπομπών, εμπορίας μάλλον ε, εκπομπών είναι μέσα στο εικόνα πολιτικής της Κίνας. Επίσης, να στηρίξουμε τον ε, διάλογο περί ενέργειας μεταξύ Ένωσης και Κίνα όσον αφορά την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας ή τη ρύθμιση αυτής. Επίσης θα μπορούσαμε να στηρίξουμε τα προγράμματα συνεργασίας για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας και βέβαια με βάση το ρυθμό των διαπραγματεύσεων για οποιαδήποτε επενδυτική συμφωνία στο μέλλον με την Κίνα θα μπορούσαμε και αυτό να το υποστηρίξουμε και αυτό παραπέμπει στα σχόλια που έκανε ο εισηγητής Ίντα σε σχέση με τα εμπορικά θέματα. Με την Ινδία, για παράδειγμα, θα μπορούσαμε μετά από το 2014, όπου ελπίζουμε πως θα έχουμε συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών με την Ινδία, θα μπορούσαμε να στηρίξουμε κάποιες πτυχές όσον αφορά ρύθμιση εμπορίου ανάμεσα στα σύνορα, ε, διάλογος ενεργειακός, ρυθμιστικό πλαίσιο, ανανεώσιμες, τέτοια πράγματα. Επίσης θα μπορούσαμε να δουλέψουμε για την πράσινη τεχνολογία και σχετικά θέματα με τρόπο ώστε να στηρίξουμε τη ερευνητική συνεργασία με την Ινδία, αλλά ίσως και πιο συγκεκριμένες εμπορικές ευκαιρίες αλλά και να προωθήσουμε προγράμματα ανταλλαγής ε, ανάμεσα σε ερευνητικά ε, Ινστιτούτα της Ευρώπης και της Ινδίας. Αυτά είναι απλά κάποια παραδείγματα που πιστεύουμε ότι εκεί θα ήταν δυνατή η στήριξη. Να τονίσω και πάλι πως είναι ένα μέσο που επιτρέπει να κάνουμε πολύ συγκεκριμένε ενέργειες για τη στήριξη συνεχιζόμενων ή μελλοντικών εμπορικών διαπραγματεύσεων με διάφορους εταίρους όταν χρειάζεται να ε, βελτιώσουμε την κατανόηση ή να προωθήσουμε την εφαρμογή ή τη συνυπογραφή μιας τέτοια συμφωνίας και όπως σα είπα αυτό το μέσο θα στηρίξει και διάφορες καινοτόμε προσεγγίσεις τις οποίες έχουμε αρχίσει να δοκιμάζουμε όπως οι τριμερείς διάλογοι η αδελφοποίηση διαφόρων σωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι τοπικών αρχών με τις αντίστοιχες άλλων χωρών, τέτοιου είδους πρωτοβουλίες. Αυτά. Θα σταθώ σε αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ κύριε Μάθιους. Παρακαλώ συνάδελφοι μην ανησυχήσετε. Είναι η πρώτη φορά ε, αυτοδιοριζόμενο προέδρο στην Επιτροπή μας, αλλά μπάση ε, πάση περιπτώσει. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Γκόλτινγκ από την ε, Δανική Προεδρία. Σας ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ καταρχήν που με καλέσατε σήμερα εδώ. Είμαι ευτυχής που βρίσκομαι εδώ και που συμμετέχω σε αυτή τη σύντομη συζήτηση. Όπως γνωρίζετε, και στο Συμβούλιο εξετάζουμε αυτή τη στιγμή αυτό το περίπλοκο πακέτο μέσων εξωτερικής δράσης, μεταξύ των οποίων είναι και αυτό εδώ, τις εταιρικές σχέσεις. Δουλεύουμε πολύ εντατικά τους τελευταίους πέντε μήνες, σχεδόν τα έχουμε καταφέρει ε, και θα μιλήσω έτσι γενικά σήμερα γιατί θα οριστικοποιηθεί η θέση μας στα τέλη του μήνα και το Συμβούλιο 26 του μηνός, Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων του 26 Ιουνίου θα εγκρίνει την θέση μας. Να σας πω λοιπόν ποια είναι η εικόνα μας ε, εμείς στην ομάδα εργασίας μας ε, έχουμε ασχοληθεί με αυτό το θέμα του μέσου εταιρική σχέσης και πιστεύω πως είναι μια πολύ καλή και περιστατωμένη πρόταση αυτή. Είναι κάτι το οποίο καλωσορίζουμε και ιδιαίτερα καλωσορίζουμε το ευρύ πεδίο εφαρμογής της ε, που ανταποκρίνεται στις πολυάριθμες ε, και πολύμορφες παγκόσμιες προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Επίσης, εξετάσαμε αυτό το μέσο για να μπορέσουμε, με στόχο να μπορέσουμε να δώσουμε στην ε, Ευρώπη του 2020 τη δυνατότητα να ανταποκριθεί ε, στις ανάγκες ανάπτυξης με αποτελεσματικό τρόπο και να μπορέσει να επιτύχει τους στόχους συνεργασίας που προκύπτουν από τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης με, τους ε, χώρες, με τις χώρες εταίρους. Πιστεύουμε ότι αυτό το μέσο θα μας επιτρέψει να το επιτύχουμε αυτό. Επίσης πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό σε αυτή τη φάση να διατηρήσουμε τη φύση αυτού του μέσου και να μην μπούμε σε υπερβολικές λεπτομέρειες περιγραφικές όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής και το είπαν ε, οι προηγούμενοι ομιλητές σε σχέση με το θέμα της ομαλής αντίδρασης και απάντησης στις ε, προκλήσεις. Και όπως το είπα και αρχικά, Επεξεργαζόμαστε την τελική μας θέση αυτή τη στιγμή και φυσικά θα καλωσορίσω τις ερωτήσεις σας, αλλά πρέπει να κατανοήσετε ότι βρισκόμαστε σε αυτή τη διαδικασία. Και έτσι θα σταθώ εδώ και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ και τώρα θα, πάρει το λόγο ο κύριος Καράνο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ που μας προσκαλέσατε σε αυτή τη συζήτηση για να συζητήσουμε δηλαδή τις μελλοντικέ προοπτικές της εξωτερικής δράσης στα πλαίσια του μεσοτερικής σχέσης. Ίσως να γνωρίζετε ότι η τράπεζά μας ήδη δρά εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει εντολή από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η οποία αναθεωρήθηκε μάλιστα πέρυσι. Έτσι έχουμε ε, το πολιτικό πλαίσιο των δραστηριοτήτων μας. Έχουμε επίσης και την εγγύηση για τις ε, δράσεις μας. Υπάρχει λοιπόν αυτό το πλαίσιο το οποίο προσφέρει καθαρές πολιτικές ενδείξεις, τι δηλαδή προσανατολισμό πρέπει να ακολουθήσουμε και συγχρόνως προσφέρει και μία εγγύηση η οποία μας επιτρέπει να δρούμε σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ αλλιώς δεν θα μπορούσαμε. Γιατί εννοείται ότι πρέπει να διατηρήσουμε το τριπλό μας α, που αποτελεί και τη βάση πάνω στην οποία δουλεύουμε. 7 δισεκατομμύρια το χρόνο δανείζουμε περίπου εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως γνωρίζετε επίσης, οι περισσότερες δραστηριότητές μας είναι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στηρίζουμε τις χώρες μέλη, ανάπτυξη και έχουμε και εταιρική σχέση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά την ε, στήριξη της πολιτικής για το 2020. Συνεργαζόμαστε στενά λοιπόν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ανάπτυξη όλων αυτών των οικονομικών ε, μέσων. Και αυτό εμπίπτει και στα πλαίσια του μεσοτερικής σχέσης. Δανείζουμε λοιπόν με μη συμβατικούς όρους καταρχήν, αλλά εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης βλέπουμε να υπάρχει η δυνατότητα να προσανατολίσουμε και εκεί τις δραστηριότητές μας, συνδυάζοντάς τες ε, με κονδύλια από τον προπολογισμό. Και αυτό έχει συμβεί τα πρόσφατα χρόνια όλο και περισσότερο με τέτοια μέσα, τα οποία μας επιτρέπουν να συνδυάζουμε τα κονδύλια με τον δανεισμό μας και τη χρηματοδότηση από άλλα βέβαια όργανα. Πράγμα που σημαίνει ότι έτσι υπάρχει πολλαπλασιαστικό φαινόμενο και πολλαπλασιάζονται ουσιαστικά τα αποτελέσματα των δράσεών μας. Το μέσο αυτό είναι πολύ αποσχόμενο για το μέλλον. Πιστεύουμε ότι πρέπει να προσθεθούν κάποια στοιχεία τα οποία να μας βοηθούν να συνδυάζουμε τους πόρους μας για την καταπολέμηση του κλίματος ή για να στηρίξουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, γιατί και εκεί έχουμε μεγάλη εμπειρία μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε εταίροι με πολλά δημοσιονομικά ιδρύματα προκειμένου να χρηματοδοτούμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Άρα εδώ πέρα υπάρχει μέλλον. 30% του δανεισμού μας περίπου εκτός της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης πηγαίνει για προσαρμογές. Κάνουμε πάντως για να κάνουμε άλλο περισσότερα σε αναπτυσσόμενες χώρες χρειαζόμαστε και και συμβατικά μέσα. Εμείς στηρίζουμε τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τις χώρες BRIC. Όταν υπάρχουν ε, εμπορικές διαφωνίες, κανονίζουμε να μην χρηματοδοτήσουμε κάποιους τομείς για να υπάρχει συνέπεια και είμαστε έτοιμοι να συμμετέχουμε στο μέσο αυτό και να δούμε πώς μπορούμε να δραστηριοποιήσουμε περισσότερα μέσα υπέρ επενδύσεων. Αυτή είναι η δικιά μας αρμοδιότητα την περίοδο 2014-2020 στα πλαίσια των ε, δημοσιονομικών προοπτικών θα έχουμε την πρόταση της Επιτροπής για την εξωτερική εντολή της ε, τράπεζά μας. Θα σας έρθει στα τέλη της χρονιάς, θα πάει και στο Συμβούλιο και ελπίζουμε και τότε να μας δοθεί ευκαιρία να συζητήσουμε για τις πολιτικές προτεραιότητες τις οποίες μπορούμε να συνεισφέρουμε μέσα στο επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο. Οι σχέσεις με χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεκινάει στη βάση συνεργασίας μεταξύ των ε, Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων, των χωρών μελών. Αυτό αποτελεί ένα καλό σημείο εκκίνησης για, τις, ε, για την αρρωγή μας και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα, σας ευχαριστώ. Πριν να ξεκινήσουμε τη συζήτηση και να δώσω και το λόγο στην συνάδελφο Μονής που το ζήτησε, και στο συνάδελφο Γκάλερ και σε όλους θα ήθελα να σας ε, ζητήσω γιατί, το εξή, γιατί στις αρχικές μου ερωτήσεις είχα υποβάλει μια πολύ συγκεκριμένη στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο και στην ε, Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Το άρθρο 5, παράγραφος 5 της πρότασης της Επιτροπής προβλέπει τη δυνατότητα δημιουργίας ενός αποθεματικού για τα μη χρησιμοποιημένα ή μάλλον μη καταχωρημένα κονδύλια γιατί αυτό να μπορεί να γίνει μόνο σε αυτό το μέσο και όχι στα υπόλοιπα μέσα, γιατί να ισχύουν διακρίσεις και πώς θα λειτουργήσει, ποιο ποσοστό κονδυλίων θα μπει εκεί και ποια θα είναι η διαδικασία για να μπουν τα κονδύλια στο αποθηματικό. Δεν ξέρω αν ανάμεσα στους προσκεκλημένους μας μπορεί κάποιος να λάβει την ευθύνη και να μου απαντήσει. Εσείς κύριε Μάθιος μήπως μπορείτε να μας απαντήσετε. Παρακαλώ. Yes, Ναι, πολύ σύντομα. Ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο. Ζητώ συγγνώμη που δεν απάντησα σε αυτή την πολύ ξεκάθαρη ερώτηση στον πρώτο γύρο των σχολείων. Πέρα από το θέμα του μεγέθους του αποθηματικού, που θα είναι μάλλον θέμα συζήτησης μεταξύ μας, ε, το, ε, ο λόγος ε, ύπαρξης του αποθέματος είναι η ίδια η ευελιξία του ίδιου του μέσου. Αν δούμε δηλαδή θέματα σε σχέση με τις προτάσεις που κάνετε για το παράρτημα. Αυτά όλα σημαίνουν δυνατότητα ταχύτατης ανταπόκρισης ή αντίδρασης στις εξελίξεις στο διεθνές προσκήνιο. Και ακριβώς γι' αυτό έχει υπάρξει αυτή η ιδέα του αποθεματικού, ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μη προβλέψιμες καταστάσεις, αλλαγές στο διεθνές περιβάλλον. Φτάνει κανείς να δει την ταχύτητα με την οποία διάφοροι συνασπισμοί έχουν αναπτυχθεί ή διαλυθεί μέσα στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για το κλίμα για να καταλάβει ότι όχι μόνο στην περίοδο του ίδιου του πολιετού δημοσιονομικού πλαισίου αλλά και μόνο μέσα σε ένα χρόνο που είναι ο συνήθις προγραμματικός μας ορίζοντας μέσα στο πλαίσιο του πολιετούς προγράμματος μπορεί να υπάρξουν αλλαγές όπου κανείς να θέλει να δαπανίσει περισσότερα χρήματα από ό,τι είχε αρχικά προβλέψει στο πουδουπού που έχει προτείνει. Όσον αφορά τον μηχανισμό, σύμφωνα με την πρόταση που έχουμε υποβάλει, ε, αυτό είναι κάτι το οποίο θα γίνει μέσω της επιτροπολογίας. Και μπορείτε να το δείτε αυτό στο κείμενο, όπως το έχουμε προτείνει. Μάλιστα. Ευχαριστώ, η κυρία Μούνης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα μιλήσω πανικά. Ανησυχώ. Ανησυχώ για αυτό το νέο μέσο. Πρώτα απ' όλα, γιατί πολύ σωστά λέτε, το γεωγραφικό εύρος είναι μεγάλο, δηλαδή περιλαμβάνονται όλες οι τρίτες χώρες. Από εκεί και πέρα μιλάμε με ασάφια, θα έλεγα, για στρατηγική σημασίας εταίρους. Και εμείς τη σκεφτόμαστε και το επανέλαβαν και όσοι πήραν το λόγο πριν, μας βάζει στο μυαλό τις χώρες BRICS, ότι πρόκειται για ένα μέσο ενίσχυσης της συνεργασίας μας και των σχέσεών μας με την Βραζιλία, την Ινδία κλπ. Εγώ πιστεύω ότι είναι σφάλμα κάτι τέτοιο. Αυτό το μέσο εταιρικής σχέσης, ναι, να έχει μεγάλο εύρος, αλλά να συμπεριλαμβάνει τρίτες χώρες που δεν εποφελούνται όμως από άλλα μέσα αρρωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης τρίτες χώρες που να μην αποφελούνται καν από άλλα μέσα θεματικά. Αν μιλάμε για στατηγική σημασία σε τότε να συμπεριλάβουμε και τις χώρες οι οποίες δεν εποφελούνται από το TCI ή άλλες χώρες οι οποίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν κοινά συμφέροντα τα οποία εμπίπτουν στις θεματικές ενότητες που καλύπτει το μέσο αυτό. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι είναι καλύτερα να μιλάμε για μεγάλο εύρος και όχι για στρατηγική σημασία σε τέρους. Γιατί η τάση είναι όλοι να έχουμε στο μυαλό μας τα BRICS, τις χώρες BRICS, πράγμα που σημαίνει ότι το περιορίζουμε αυτό το μέσο εταιρική σχέση. Δεύτερον, εδώ που βρισκόμαστε τώρα με τα διάφορα οικονομικά μέσα και τις αλλαγές που γίνονται πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί με το συντονισμό μεταξύ τους. Το DCI που είναι για την συνεργασία για την ανάπτυξη αναφέρεται στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι το 90% των κονδυλίων του μέσου αυτού απευθύνονται σε προγραμματισμό, προγράμματα κτλ. που σέβονται τις αρχές της ε, επίσημης αναπτυξιακής αρρωγής. Χρησιμοποιείται δηλαδή όμως πέρα από τα πλαίσια αυτής της αρρωγής. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν με το 10% που υπάρχει στο μέσο ανάπτυξης. Δεν πρέπει να το βάλουμε στο μέσο της συνεργασίας με τρίτες χώρες δηλαδή το DCI πρέπει να τηρεί τους όρους του ΚΑΤ που πρόκειται για την επίσημη αναπτυξιακή αρρωγή δηλαδή. Συνεπώς, με τέτοιους όρους, ώστε μέσω ενός μέσου συνεργασίας με τρίτες χώρες να προχωρήσει και όχι με προγράμματα τα οποία δεν έχουν καμιά σχέση με την ανάπτυξη. Δηλαδή δεν βλέπω γιατί με το μέσο αναπτυξιακής ε, ε, βοήθειας, να χρηματοδοτούμε ε, προγράμματα τα οποία δεν έχουν καμιά σχέση με την ανάπτυξη, ενώ υπάρχει άλλο μέσο το οποίο μπορεί να συμπεριλάβει και αναπτυσσόμενες χώρες για προγράμματα τα οποία δεν έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη. Το ίδιο θα έλεγα και για το μέσο για την πυρηνική ασφάλεια. Υπάρχει ένα τέτοιο μέσο και σε αυτό εδώ το μέσο για τρίτες χώρες αναφέρεται στις θεματικές αρμοδιότητες και η πυρηνική ασφάλεια. Ναι, αλλά πρέπει να δούμε το κάθε μέσο τι μπορεί να χρηματοδοτήσει και τι όχι. Να μην υπάρχουν επικαλύψεις όταν μιλάμε για την πυρηνική ασφάλεια, ε, να χρηματοδοτηθεί αυτή από το δικό μέσο για την πυρηνική ασφάλεια και όχι από άλλα. Έπειτα πρέπει να υπάρχει μεγάλη διαφάνεια και να ε, υπάρχει και κάποια ευελιξία για αυτό το μέσο. Οτιδήποτε έχει να κάνει με σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τρίτες χώρες και έχει να κάνει και με τη στρατηγική 2020 στην εξωτερική της διάσταση, με τα αμοιβαία συμφέροντα Ευρωπαϊκής Ένωσης και οποιαδήποτε άλλες τρίτες χώρες. Αλλά δεν συμπεριλαμβάνεται στα άλλα μέσα, τότε ναι, να συμπεριληφθεί εδώ. Γι' αυτό μιλάμε για ευελιξία. Αυτήν θέλει να διατηρήσει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μίλησα πριν για τις χώρες BRICS. Υπάρχουν άλλα μέσα που οριοθετούνται ή δεν οριοθετούνται γεωγραφικά. Γι' αυτό λέω ε, να μην μιλάμε για στρατηγική σημασία τέρους. Και υπάρχει και η έκθεση Μπροκ που μιλάει για αυτά, που αναφέρεται στην ε, εξωτερική πολιτική και λέει ότι καλωσορίζουμε αυτό το νέο μέσο για τους ε, εταίρους μας στρατηγική σημασία. Μα όχι, αν βάλουμε εταίρους στρατηγική σημασία να βάλουμε και άλλους. Μην δημιουργούμε με αυτόν τον τρόπο ένα μέσο, το οποίο τελικά θα εξυπηρετήσει, θα ενισχύσει τέλο πάντων τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης μόνο με τις χώρες BRICS. Η κάθε χώρα να είναι στη θέση της. Οι σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανάλογα με το πόσο στενές είναι, περιλαμβάνονται στο ένα ή στο άλλο μέσο, σε αυτό ή σε άλλο. Αλλά να ξέρουμε γιατί πράγμα μιλάμε κάθε φορά. Κατά τα άλλα, κύριε Μάουρο, πιστεύω ότι η έκθεσή σας επικεντρώνεται σωστά. Ίσως να αναφέρονται υπερβολικά η G7, η G20 και λίγο οι διαπεριφερειακές σχέσεις μεταξύ των δικαιούχων χωρών. Αλλά κατά τα άλλα εντάξει. Αυτό που δεν μας αρέσει τόσο πολύ είναι πώς βλέπει το θέμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω πως συμμεριζόμαστε και την ε, θέση για περαιτέρω διεύρυνση από τις χώρες BRICS. Ο συνάδελφος Γκάλερ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ είμαι ευνοϊκά διακείμενος απέναντι σε αυτή την πρόταση για αυτό το νέο ε, μέσο γιατί θεωρώ πως το χρειαζόμαστε και ότι λείπει. Το έχουν πει συχνά οι συνάδελφοι, ότι συχνά γίνεται μια, ένας αγώνας για το μέσο συνεργασίας ε, και για την ανάπτυξη και ε, προσπαθούμε να βοηθήσουμε αυτές τις χώρες, αλλά όσον αφορά το ICI ή το ICI είναι συχνά υπάρχουν ε, δυσκολίες στην χρήση του ή στην εφαρμογή, στην εφαρμογή του. Τώρα, ε, τούτο εδώ είναι ένα ε, μέσο το οποίο δεν έχει βασικό στόχο να βοηθήσει τις ε, τρίτες χώρες, αλλά λαμβάνει μόνο, αλλά να λαμβάνει υπόψη και τα δικά μας συμφέροντα, τα οποία ταυτόχρονα μπορεί να ενισχύσουν και τη συνεργασία. Αυτή λοιπόν την ευελιξία την βλέπουμε και στην παράγραφο 2, μάλλον άρθρο 2, παράγραφο 2. Δηλαδή να στηρίξουμε κυρίως μέτρα συνεργασίας με τις αναπτυσσόμενες χώρες που παίζουν σημαντικό ρόλο. Γίνεται λόγος δηλαδή για αναπτυσσόμενες χώρες καταρχήν. Δηλαδή υπάρχει μια ευελιξία. Ε, πιστεύω και ελπίζω ότι αυτή η ευελιξία δεν αφορά μόνο τις χώρες αλλά και την εφαρμογή στην, στο, μέσο αυτού. Η τροπολογία δηλαδή όπου λέει ότι αντί να έχουμε ενδεικτικά πολιτή προγράμματα θα έχουμε ένα τέτοιο έγγραφο το οποίο θα είναι το μέσο του στρατηγικού προγραμματισμού. Αλλά εδώ τι χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε, όπως ε, λέει και στο 6 και στο 7, όπου χρειάζονται μικρές ε, τροποποιήσεις, όπως ε, η πρόταση που γίνεται μέσω της τροπολογίας και δίνεται έτσι μεγαλύτερη ευελιξία. Διότι εδώ το θέμα δεν είναι να τα, να τα ε, προγραμματίζουμε όλα ιδιαίτερα γραφειοκρατικά. Χρειάζεται μεγαλύτερη ευελιξία και γι' αυτό στα πλαίσια της δημιουργίας Θα ήμουν λοιπόν διατεθειμένος να δώσω δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Κομισιόν να αντιδράσουν ε, με βάση τι χρειάζεται στις διάφορες χώρες. Ανέφερε η συνάδελφος ε, Μουνίθ την, ε, τις χώρες BRIC. Υπάρχουν και άλλες χώρες όπου θεωρώ ότι μπορούμε να αναπτύξουμε συγκεκριμένα προγράμματα. Βεβαίως θα παίξουν ρόλο οι χώρες BRIC, ενδεχομένω και εξέχοντα ρόλο, αλλά κατά κανένα τρόπο δεν πρέπει να περιορίσουμε ε, το πεδίο εφαρμογή αυτού του μέσου μόνο σε αυτές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τάνοκ. Ευχαριστώ. Δυστυχώς ε, ε, τα έχουμε ανακατέψει όλα, έχουμε τόσο πολλά μέσα και για μας τους καημένους, τους βουλευτές ε, ούτε να τα θυμηθούμε δεν μπορούμε και αλλάζουν και όνομα. Ίσως επίτηδες για να μην καταλαβαίνει ο κοινό άνθρωπος περί τίνος πρόκειται. Από ό,τι το καταλαβαίνω εγώ και η ομάδα μου, αυτό το νέο μέσο για τη συνεργασία από πρώτη άποψη μοιάζει να έχει καλές προθέσεις να στηρίξουμε με πιο ευέλικτο τρόπο οικονομικά αυτά τα μεγάλα σφαιρικά θέματα όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να παίξει ρόλο βασικό να είναι περίπου ισότιμος με το G8 της BRIC. Ξέρετε ότι αυτό είναι επίμαχο πολύ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι διμερείς συμφωνίες με μεγάλες ε, ε, χώρες όπως η Ινδία και η Κίνα ξέρετε ότι έχουν αποσυρθεί. Για ποιο λόγο να δίνουμε βοήθειες σε αυτές τις χώρες με τέτοιες διαστάσεις, αλλά είμαστε επιφλακτικοί ως ομάδα για το κατά πόσον ε, υπάρχει προστιθέμενη αξία μέσω χρήσης αυτού του νέου μέσου. Έχω ανησυχίες για το πώς θα επιτηρείται το μέσο αυτό, πώς θα υπάρχει ανεξάρτητος λογιστικός έλεγχος για να δούμε την προστιθέμενη αξία, τις προτεραιότητες, ε, μέσω των οποίων θα χρηματοδοτούνται προγράμματα πέρα και πάνω από όλα όσα διμερώς ήδη πράττουν τα κράτη-μέλη έναντι των BRIC και μεταξύ διαφορών άλλων ε, κυρίων παραγόντων στρατηγικών εταίρων. Και τι προστιθεμένη αξία. Μιλήσαμε για την καταπολέμηση της ε, κλιματικής αλλαγής, βεβαίως σημαντικό θέμα, αλλά ήδη υπάρχουν μια σειρά διεθνείς πρωτοβουλίες στα πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών. Γιατί χρειάζεται και κοινοτική παρέμβαση χωριστά από όσα κάνει ο Οργανισμός Ομένων Εθνών. Επίσης, λόγω της σοβαρής λιτότητας στα κράτη-μέλη, λόγω της υπαρξιακής κρίσης της Ένωσης, των προβλημάτων που έχει η Ισπανία με την ανακεφαλαιοποίηση των ε, τραπεζών, γιατί να δώσουμε πάνω από ένα δις στο πλαίσιο των πολιετών ε, προοπτικών για τα επόμενα δηλαδή 7 χρόνια τεράστια ανάπτυξη σε σχέση με την προηγούμενη χρηματοδότηση που ήταν μόνο 200 εκατομμύρια. Από πού θα βγουν όλα αυτά τα επιπλέον χρήματα. Εντάξει, με καθησυχάζει κάπως ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων που γενικά λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες της αγοράς μοιάζει να το υποστηρίζει. Επίσης, με καθησυχάζει το ότι αντιτίθεται οι σοσιαλιστές. Άρα καλό πράγμα θα είναι. Ιδιαίτερα για θέματα όπως η πυρηνική ενέργεια και η πυρηνική ασφάλεια που την υποστηρίζει η ομάδα μου. Βεβαίως για την αναπτυξιακή βοήθεια εγώ έχω υπάρξει ε, ε, υπέρμαχος της βοήθειας προς το κέρας της Αφρικής και την ε, νέα αυτή χώρα που λέγεται Σομάλιλάντ ε, αυτή η νέα χώρα, το Σομάλιλαντ, θέλει να φτιάξει φυλακές για να κλείσει κάποιος από τους πειρατές. Ε, και όμως δεν μπορεί να ληφθεί αρκετή χρηματοδότηση λόγω των περιορισμών των μέσων αναπτυξιακής βοήθειας. Άρα θα ήταν σκόπιμο να υπάρξουν αυτές οι βοήθειες για να διαχωρίσουμε τους ε, κοινού εγκληματίες αυτές τις φυλακές από τους πειρατές. Τώρα δεν είναι δυνατόν. Οι νόμοι τώρα για την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια είναι τόσο περιοριστικοί που δεν το επιτρέπουν. Ίσως λοιπόν θα μπορούσαμε να χρηματοδοτήσουμε κάπως και κάποια θέματα ασφάλειας μέσω συγκεκριμένων προγραμμάτων για τη διεθνή συνεργασία για την ασφάλεια στον Ινδικό ωκεανό μέσω και των προγραμμάτων Αταλάντα και Unifor. Να δούμε λοιπόν τι ανάγκες θα πρέπει να ε, χρηματοδοτήσουμε. Έχει η ομάδα μου ακόμη κάποιε επιφυλάξει, αλλά νομίζω ότι είναι καλέ οι προθέσει του και ίσω είναι αναγκαίο αυτό το νέο μέσο. Αλλά η ομάδα μου επιφυλάσσεται όσον αφορά τη στάση τη στην τελική ψηφοφορία, μέχρι να το μελετήσουμε λίγο ακόμη, ε, συζητώντα με τι κυβερνήσει και του εμπειρογνώμονε για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Εάν δεν υπάρχουν άλλοι συνάδελφοι που να θέλουν τον λόγο, πριν να δώσω το λόγο στους ε, καλεσμένους μας, θα ήθελα να ρωτήσω την κυρία Ανδρικένε αν έχει περαιτέρω σχόλια να κάνει, αν θεωρεί ότι είναι ικανοποιητικέ οι απαντήσεις που έλαβε. Σας ευχαριστώ. Εκτιμώ πραγματικά τις απαντήσεις που έλαβα στις ερωτήσεις που, που έθεσα, εκτός από μία το ερώτημά μου του μεριδίου 20% ε, για την, τα μη καταχωρημένα κονδύλια. Παρακαλώ να το απαντήσετε και έπειτα για να ολοκληρώσω αυτό που έλεγα νωρίτερα, ότι δηλαδή Πιστεύω πως είναι πολύ σημαντικό το, οι συνομοθέτες, το Ευρωκοινοβούλιο και το Συμβούλιο, να συμμετέχουν ε, το ίδιο στην ε, λήψη στρατηγικών αποφάσεων. Και γι' αυτό στην έκθεσή μου προτείνω ενδεικτικές τομείς συνεργασίας και κατανομής οικονομικής και τροποποίησης ότι θα πρέπει να είναι ε, αντικείμενα κατεξουσιοδότησης πράξεων. Κατεξουσιοδότηση πράξεων και η στρατηγική 2020 επίσης να περιλαμβάνεται σε αυτή τη στρατηγική, την νομοθεσία και τη στρατηγική. Δεν θέλω περισσότερες απαντήσεις, θα ήθελα απλά οι συνάδελφοι από την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και την Κομισιό να το λάβουν αυτό υπόψη. Σας ευχαριστώ πολύ και τώρα το λόγο έχουν οι προσκεκλημένοι μας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω στην κυρία Μούνης. Ε, νομίζω πως υπάρχει κάποια παρεξήγηση. Αυτό το μέσο θα πρέπει και θα έχει παγκόσμια εμβέλεια. Δηλαδή δεν είναι μόνο για τις χώρες BRICS. Είναι για όλες αυτές τις χώρες όπου θα ήταν προς, ε, που θα ήταν ενδιαφέρον για, σε κάποια φάση χρονική για την Ευρωπαϊκή Ένωση να ξεκινήσει κάποια προγράμματα. Σαφώς δηλαδή είναι σχεδιασμένο ώστε να καλύψει ολόκληρο τον κόσμο δυνητικά. Βέβαια ε, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι ζητάμε ένα σχετικά περιορισμένο ποσό κονδύλι 153 εκατομμύρια ευρώ το ετησίως για μια περίοδο 7 ετών. Δεν είναι και πολλά χρήματα αν σκεφτείτε ότι πρέπει να καλυφθεί ολόκληρος ο κόσμος και γι' αυτό και χρειάζεται να έχουμε και κάποιους γενικούς προσανατολισμούς. Και αυτό είναι κάτι που θέλω να πω απαντώντας και στο πόσο τελικά τι κερδίζουμε από αυτό εδώ το πρόγραμμα. Το μέσο αυτό θα χρησιμοποιηθεί ως μόχλευση, ως μοχλός. Δεν χρειαζόμαστε τόσα πολλά χρήματα, αλλά θέλουμε αυτά τα χρήματα να χρησιμοποιηθούν με ευέλικτο τρόπο σε συνδυασμό, όποτε αυτό είναι δυνατό, με τα όσα είπε ο συνάδελφος από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Έτσι ώστε δηλαδή να έχουμε περισσότερη, από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, με συγχωρείτε, ώστε να έχουμε δηλαδή πολύ πιο μεγάλο αντίκτυπο στην πραγματικότητα. Αν δείτε τι έκανε το ICI και το ICI SIN, μόνο 17 χώρες κάλυπταν. Εδώ μιλάμε για ένα μέσο, ε, όπως είπαμε, παγκοσμίου εμβέλειας και Φυσικά θα προσπαθήσουμε να εξασφαλίσουμε την παραπληρωματικότητα με τα άλλα δημοσιονομικά μέσα, ιδιαίτερα με το μέσο για την πυρνική ενέργεια που αναφέρατε και, και άλλα μέσα όπως το DCI. Θα ήθελα λοιπόν ο, ο συνάδελφος, αν επιτρέπεται ο κ. Μάθιου Έλλης, να μπορέσει έτσι να απαντήσει σε άλλες ερωτήσεις που έθεσαν οι προβλεφτές. Παρακαλώ, κυρία Μάθιους. Σας ευχαριστώ που μου ξαναδίνετε το λόγο. Αυτό που τονίστηκε και δεν καλύψαμε ικανοποιητικά ήταν το θέμα της ευελιξίας σύμφωνα με το άρθρο 5 της πρότασής μας. Αυτό που θα ήθελα να πω από αυτό είναι το εξής και πάλι μεταξύ λογικών ανθρώπων μπορούμε να συζητήσουμε για το ποιο θα είναι το κατόφλι για μια τέτοια μη σημαντική αλλαγή ή τροποποίηση. Πάντως η ιδέα είναι ε, εκεί με το στόχο ενός ε, σταθερού προγράμματος. Ε, δεν μιλάμε για την εισαγωγή ιδεών που δεν έχουν προηγουμένως συμφωνηθεί. Η ιδέα είναι ότι έχουμε ένα πολιετές πρόγραμμα που μπορεί να διαρκέσει 3-4 χρόνια, αν δούμε και την περίοδο του πολιετούς δημοσιονομικού προγράμματος, να μπορούμε δηλαδή να μετακινήσουμε χρήματα ανάμεσα στις προτεραιότητες μέσα στο πλαίσιο του προγραμματισμού. Αυτό θα γίνεται με προσαρμογές ετήσιες μέσα στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος. Γι' αυτό έχει σχεδιαστεί, να μπορούν να μετακινηθούν χρήματα ανάμεσα σε ήδη συμπεφωνημένε προτεραιότητε. Συμβαίνει στο πλαίσιο κάποιων προγραμμάτων. Άμα δεν λειτουργήσουν ε, τελικά ε, και δεν θα πρέπει να τους δώσουμε άλλα χρήματα μέσα στο πλαίσιο, το γενικό, το κονδύλι που έχει αρχικά συμφωνηθεί. Αυτό είναι ο στόχο αυτού του αποθέματο. Πρέγω, ah, Yes, uh, thank you. Uh. Ευχαριστώ. Να συμπληρώσω σε σχέση με αυτά που είπε η κυρία Μουνίθ για τους στρατηγικούς εταίρους BRIC και τα λοιπά. Όπως ε, ήδη υπόθηκε. Βεβαίως θα είναι παγκόσμια η κάλυψη. Αλλά οι πιστώσεις ε, στη διάθεσή μας δεν μας επιτρέπουν να μην καθορίσουμε προτεραιότητες. Έστω ενδεικτικές για Κοινοβούλιο και Συμβούλιο. Αλλά παγκόσμια κάλυψη δεν σημαίνει μόνο στρατηγική εταίρη ότι θα χρηματοδοτήσουμε μόνο στρατηγικού εταίρους. Θα χρηματοδοτήσουμε συμπληρωματικά με τα άλλα μέσα διάφορες δραστηριότητες. Μιλάτε για δραστηριότητες ε, διμερούς βοήθειας, αναπτυξιακής βοήθειας. Εκτός λοιπόν από τις διμερείς υπάρχει βεβαίως κάποια ευελιξία λοιπόν στα περιφερειακά και τομεακά προγράμματα του νέου κανονισμού για την αναπτυξιακή βοήθεια που επιτρέπουν τη χρηματοδότηση περιφερειακής βοήθειας στη Λατινική Αμερική. Αυτό λοιπόν το νέο εταιρικό μέσο μπορεί να συνδυαστεί με άλλα μέσα χρηματοδότησης. Θα μας επιτρέψει να χρηματοδοτήσουμε προγράμματα στη Λατινική Αμερική. Το μέσο για την πυρηνική ασφάλεια με τον ίδιο τρόπο θα αξιοποιηθεί. Έχει πολύ συγκεκριμένο στόχο στα πλαίσια της συνθήκης Ευρατόμ. Θα λειτουργήσει λοιπόν κάπως διαφορετικά, γιατί λειτουργεί διαφορετικά η συνθήκη Ευρατόμ από ότι αυτό το μέσο. Υπάρχει λοιπόν η δυνατότητα να βοηθήσουμε τις χώρες να βελτιώσουν την ασφάλεια των πυρηνικών τους εγκαταστάσεων για την παραγωγή ενέργειας. Γιατί είναι προς το συμφέρον μας. Ξέρετε, όταν υπήρξε ατομικό δυστύχημα στην Ιαπωνία, έχει παγκόσμιες επιπτώσεις. Είχε παγκόσμιες επιπτώσεις. Ο κύριος Τάνοκ μίλησε για την καταπολέμηση της πειρατείας στο κέρα της Αφρικής. Μα υπάρχει ήδη ένα όργανο που καλύπτει αυτή τη δραστηριότητα. Και φυσικά, στην πρόταση προς την αρχή επί του προϋπολογισμού περιλαμβάνεται η χρηματοδότηση αυτή τη δραστηριότητα. Δεν πρόκειται για επικάλυψη, αλλά για συμπληρωματικότητα. Αυτό μπορεί να προσφέρει αυτό το νέο μέσο που έχει, όπω είπαμε, παγκόσμια εμβέλεια. Οπότε επαναρχόμεθα στο πρώτο σημείο. Είναι πολιτικό μέσο. Όχι για αναπτυξιακή βοήθεια, αλλά για την προώθηση των πολιτικών της Ένωσης και των ε, νέων στρατηγικών μας. Αναφέρθηκε ήδη από τον εισηγητή ότι εντάσσεται στα πλαίσια του Ευρώπη 2020. Ευχαριστώ. Ο κύριος Καράνο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Καταληκτικά, κατά τη γνώμη μας, οπωσδήποτε αυτό το μέσο θα επιχειρήσει να αυξήσει την αποδοτικότητα και όλων των άλλων μέσων της Ένωσης φυσικά και των μέσων της τράπεζάς μας. Έτσι θα έχουμε υψηλότερη πολιτική και οικονομική μόχλευση. Ο συνδυασμός αυτών των ε, σχετικά περιορισμένων ε, ποσών, όσο και αν αυξάνεται με αυτό το νέο μέσο, για 7 χρόνια για όλες ε, τις χώρες, τις, όλες τις τρίτες χώρες, είναι περιορισμένο. Θα έχουμε λοιπόν υψηλότερες επιπτώσεις. συνδυάζοντας για παράδειγμα δάνεια με επιδοτήσεις. Αλλά επιδοτήσεις όχι μόνο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιδοτήσεις που στην ουσία θα είναι συγχρηματοδοτήσεις για το κοινό καλό. Θα συμβάλλουν δηλαδή και οι χώρες αυτές. Πρέπει να το διερευνήσουμε στο μέλλον περισσότερο αυτό. Όπως ξέρετε δεν χρησιμοποιούμε για την δανειοδότηση χρήματα φορολογουμένων. Δανειζόμαστε από τις αγορές. Πέρυσι περίπου 76 δις. 40-50% των ε, ποσών αυτών προέρχονται από μη Ευρωπαίους επενδυτές και 90% πηγαίνει στα κράτη-μέλη. Και ίσως να χρειαστεί να πάνε και περισσότερα λόγω της κρίσης. Είναι σημαντικό λοιπόν να υπάρχει εταιρική σχέση με μη ευρωπαϊκές ε, χώρες που είναι στρατηγικοί εταίροι μας. Γιατί αυτό συμβάλλει και στη δική μας χρηματοδότηση. Ευχαριστώ. Η Προεδρία. Η Δανέζικη Προεδρία. Κάποια σχόλια. Νομίζω ότι πολλοί παρεμβαίνοντε εξέφρασαν τις ίδιε ανησυχίες που εκφράστηκαν και στο Συμβούλιο, στις ομάδες εργασίας όταν συζητάμε για το θέμα αυτό. Κοινέ λοιπόν είναι οι ανησυχίε μας. Πιστεύω ότι στη συνέχεια, στον τριμερή διάλογο, θα καταλήξουμε σε κοινού παρονομαστές. Για αυτό το μέσο που διαμακρών ε, παρουσίασαν οι συνάδελφοί μου εξ αριστερών μου, προέκυψε ότι πρέπει να διασφαλίσουμε την αποφυγή επικάλυψης. Υπάρχουν πολλά ή εφτά μπορούν να αφορούν ε, τον ίδιο τομέα, την ίδια περιοχή. Φυσικά πρέπει να αποφύγουμε τις πατάλες. Να υπάρχει τριπλή και τετραπλή επικάλυψη μέσω τριών ή τεσσάρων διαφορετικών μέσων δηλαδή. Είναι βασικό αυτό. Να υπάρχει σωστή συμπληρωματικότητα μεταξύ αυτού του νέου μέσου και των άλλων μέσων που έχουμε. Το τόνισαν ε, πολλοί παρεβαίνοντες ε, και είναι σημαντικό. Βεβαίως προσβλέπουμε ιδιαίτερα και στη συνέχιση της διαδικασίας. Ξέρω ότι θα υποβάλλετε συντόμως τροπολογίες και το Συμβούλιο θα ε, τις εξετάσει προσεχώς μέσα τον Ιούνιο θα προχωρήσουμε λοιπόν. Ευχαριστώ τον Πρόεδρο Μπροκ. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ που είχα αυτήν την θαυμάσια εμπειρία να προεδρεύσω για μια ώρα. Το επόμενο ε, θέμα είναι η Αλγερία. Παρακαλώ όλοι οι εκπρόσωποι ε, τρίτων οργάνων, οι καλεσμένοι και οι δημοσιογράφοι παρακαλούνται να αποχωρήσουν πριν ξεκινήσουμε τη συζήτηση για το θέμα αυτό. Γιατί θα γίνει και